Υποτίθεται ότι μόνο προσωρινά και ως ίστατο μέσο επιτρέπονται ε, οι εσωτερικοί συνοριακοί ε, έλεγχοι, αλλά επανεισάγονται από τα κράτη-μέλη ε, αυθαίρετα. 50 φορές έχουν παραταθεί τέτοιοι έλεγχοι, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει επιβάλει ποινές στι χώρες αυτές. Φέτος, τον Απρίλιο, η Γερμανία παρέτεινε για άλλη μία φορά τους ελέγχους στα σύνορα με την ε, Αυστρία. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν ε, όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ε, αντιδρά είμαι πολύ περήφανη για το ψήφισμα του Κοινοβουλίου. Για να υπερασπιστούμε την ελεύθερη κινητικότητα ελπίζω να υπερψηφιστεί το ψήφισμα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Κολάκουση, ένα λεπτό. Αγαπητοί συνάδελφοι, η ισοτιμία, η πολυγλωσία και τα κοινά σύνορα είναι από τα θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε στην πανδημία COVID-19 να διατηρεί μια παράδοξη κατάσταση όπου τέσσερις χώρες που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να βρίσκονται στο χώρο Σέγγεν, ενώ τέσσερι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ρουμανία, η Βουλγαρία, η Μάλτα και η Κροατία, που είναι εδώ πολλά χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, είναι εκτός του χώρου Σέγγεν. Θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε, να μην φυστούμε προσπαθειών, ώστε από φέτο και όλα και οι τέσσερις υπόλοιπε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μπουν στο χώρο Σέγγεν και να μην επιτρέψουμε το κλείσιμο των συνόρων όπως είχαμε τον τελευταίο καιρό, όπου με χώρες επανέφεραν τους συνοριακούς ελέγχους ε, συνταράσσοντας από ε, θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι ε, ένας χώρος χωρίς σύνορα, ένας κοινό χώρος για όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Πόκνταν για ένα λεπτό. Κυρίε και κύριοι, η συμπερίληψη της Ρουμανίας στον χώρο Σέγγεν δεν είναι κάτι α, τυπικό και διαπιστώνω ότι η μοναδική σχέση που έχει η Ρουμανία με τον χώρο Σέγγεν είναι ότι χορηγούμε ε, εποχιακούς εργαζόμενους αλλά δεν έχουμε το ίδιο καθεστώς ε, που έχουν άλλα κρατημέλη και άλλοι εργαζόμενοι από τα άλλα κρατημέλη σε ό,τι αφορά την ε, υγειονομική περίθαλψη και το καθεξή. Και συνεχίζεται να μπλοκάρεται η είσοδο τη Ρουμανία στο Σέγγεν παρά το γεγονό ότι πληρούνται οι τεχνικοί όροι οι τεχνικές διατάξεις. Χρειαζόμαστε λοιπόν ε, ευρωαισιοδοξία. Μιλάμε σήμερα για μια λειτουργική, ένα λειτουργικό χώρο Σέγγεν. Δεν τον ενδυναμώνουμε όμως. Και αυτό το τονίζουμε. Γιατί βλέπουμε ότι και η Ολλανδία και άλλοι είναι κατά της εισόδου της Ρωμανίας εδώ και χρόνια, χωρίς ε, λόγο. Η Ρουμανία έχει κυβέρνηση από πλευρά της ΕΛΚΑ. Γιατί λοιπόν μπλοκάρετε η είσοδο της ε, Ρουμανίας. Δεν το καταλαβαίνουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ λέει ο Πέρδο, και τώρα το λόγο έχει η κυρία Σίπελ. Για ένα λεπτό. Έχετε το λόγο. Ε, ευχαριστώ. 35 χρόνια Σέγγεν. Μια πραγματική επιτυχία. Απίστευτη. Και έρχεται μετά η πανδημία και με το που κλείνουν τα σύνορα φαίνεται ότι το Σέγγεν δεν είναι κάτι το αυτονόητο. Είναι όμως απαραίτητο, αναπόσπαστο σημείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πραγματικά κάτι απαραίτητο για τη διακίνηση αγαθών, προϊόντων, φαρμάκων και άλλων ε, ζητημάτων. Αλλά και πολλά παραπάνω περιλαμβάνει ο χώρος Σέγγεν. Την καθημερινή ζωή και ελεύθερη μετακίνηση των ε, ανθρώπων που μένουν κοντά στα σύνορα. Πρόκειται για το θεμελιώδη Δηλαδή αρχή της κατανόησης, αλληλοκατανόησης και της υπέρβασης των διαφορών που έχουμε. Γι' αυτό λοιπόν καλό την Κομισιόν, το Συμβούλιο και τα κράτη-μέλη να ενισχύσουν το χώρο Σέγγεν και να μας επιτρέψουν να ζήσουμε σε καθημερινό επίπεδο την Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, λέει και Πρόεδρος. Κέλλερ, για ένα λεπτό. Κυρία Επίτροπε, Αγαπητή Ιλβα Γιώχανσον, στην ε, αρχή της πανδημίας COVID-19 η Ευρώπη κατακαιρματίστηκε. Τα περισσότερα κράτη-μέρη επανέφεραν τους, ε, τους ελέγχους στα σύνορα και έτσι χιλιάδες πολίτες, διασυνοριακά εργαζόμενοι, οικογένειες ε, μπλοκαρίστηκαν, έμειναν χωριστά και το βίωσα και εγώ γιατί ε, είμαι κάτοικος Στρασβούργου, μιας ε, πόλης κοντά στα σύνορα. Ήταν πραγματικά ενίκουστη και πρωτοφανής αυτή η κατάσταση. Θα ήθελα λοιπόν να οργανώσουμε πριν το καλοκαίρι ένα ε, restart, μια επαναφορά της και ανάλυση της κατάστασης για να δούμε πώς θα μπορούσαμε να είχαμε αντιδράσει καλύτερα και να δώσουμε κάποιες λειτουργικές λύσεις και απευθύνω έκκληση σε όλου του συναδέλφου για έναν πιο ολοκληρωμένο μηχανισμό διαχείριση των συνόρων μα. Θα σα πρότεινα λοιπόν να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε νέα απειλή στην ελεύθερη διακίνηση ιδιαίτερα σε περίπτωση δεύτερου κύματο τη πανδημία. Όπω μα υπενθύμησε ο πρόεδρο Λόπε Ακυλάρ, η ελεύθερη διακίνηση είναι νευραλγικός παράγοντας και για την οικονομία μας και για την απασχόληση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κυρία Κελέρ. Το λόγο έχει τώρα ο κύριος Ερικ Μάρκαρτ. Για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Δύσκολους καιρούς ζούμε και ιδιαίτερα σε τέτοιους καιρούς είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τι ευτυχία είναι να ζούμε αυτήν την εποχή στην Ευρώπη. Φανταστείτε να είχαμε γεννηθεί πριν 100 χρόνια. 50 εκατομμύρια νεκροί από την Ισπανική γρήπη μόλις είχε τελειώσει ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, η οικονομική κρίση ε, και κατόπιν ήρθαν οι Ναζί στη Γερμανία που οδήγησαν στο χείλος του γκρεμού όλον τον κόσμο. μετά το τέλος του πολέμου ε, ε, Λίγα χρόνια μετά χτίστηκε το τείχος του Βερολίνου που δίχασε στα δύο την Ήπειρό μας. Ιδιαίτερα σε τέτοιες ε, εποχές κρίσης είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τι έχουμε πετύχει και να βρούμε στοχευμένα μέτρα για να καταπολεμήσουμε τον ιό και όχι ε, το ευρωπαϊκό εγχείρημα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Τζαμπάς, και ένα λεπτό. Ε, Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, καταρχήν θα ήθελα να διορθώσω τους συναδέλφους που ισχυρίστηκαν ότι τα κράτη-μέλη έκαναν λάθος με την επαναφορά των, σύνορων, των ελέγχων στα σύνορα. Όχι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν αυτή που απέτυχε σε θέματα ελέγχου των σύνορων. Ήταν τελείω ανεπαρκή η συμπεριφορά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανάγκασε τα κράτη-μέλη σε μονομερεί λύσει και μέτρα. Για να έχουμε ασφαλή εσωτερικά σύνορα, θα πρέπει να έχουμε πρώτα ασφαλή εξωτερικά σύνορα. Είναι αδύνατο να έχουμε εκατομμύρια μετανάστες που εισέρχονται χωρίς πρόβλημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ταυτόχρονα θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και το θέμα της εσωτερικής ασφάλειας. Αυτό είναι αδύνατο και μας το έδειξε για μία ακόμη φορά η πανδημία COVID-19. Θα πρέπει επίση να προσθέσουμε και την τελείω ανεύθυνη συμπεριφορά κάποιων χωρών, όπω οι κάτω χώρε, που μπλοκάρουν την είσοδο τη Βουλγαρίας και Ρουμανία στο χώρο Σέγγεν. Αυτό είναι απαράδεκτο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και τώρα το λόγο έχει για ένα λεπτό η κυρία Μπιόρκ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Όταν συζητάμε το Σέγγεν δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι δεν είναι μόνο θέμα ελεύθερης κινητικότητας εντός ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και να μπορούμε να κάνουμε διακοπές ε, χωρίς το διαβατήριο στην τσέπη μας. Το Σέγγεν συνδέεται και με το κλείσιμο των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τώρα αυτό έχει φτάσει σε επίπεδα τρομακτικά. Το βλέπουμε στα σύνορα της Ελλάδας, το βλέπουμε στα Βαλκάνια. Βλέπουμε μια πολιτική που βάζει πάνω από την προστασία των ανθρώπων την προστασία των, των εξωτερικών συνόρων. Δεν μπορούν ναι, όμως οι ελευθερίες μας να βασίζονται σε θηριωδίες στα εξωτερικά ε, σύνορα. Και δυστυχώς ένα ε, τέτοιο χτυπητό παράδειγμα είναι η χώρα της Προεδρίας, η Κροατία, όπου ε, βλέπουμε παράνομη επαναπρόθεση επανειλημμένα από πλευράς της αστυνομίας. Θα πρέπει να δεν επιτρέπεται να επιβραβεύουμε μία χώρα όταν ε, παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει η κυρία Ντουιπών για ένα λεπτό. Ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, κυρία Επίτροπε, τριών ετών ήμουν όταν έπεσε το τείχος του Βερολίνου, δεκατριών ήμουν όταν ε, μπήκε στη συνθήκη του Άμστερντα με το Σέγγεν και η Ευρώπη πάντα ήταν μέρος της ζωής μου. Εγώ έχω ζήσει την Ευρώπη ως ανοιχτή και ελεύθερη ήπειρο και ειλικρινά ποτέ δεν περίμενα να ξαναδώ συνοριακούς ελέγχους. Καταλαβαίνω ότι λόγω της φύσης της πανδημίας και Τη ε, ισχυωστής ε, το να κλείσουμε τα σύνορα χωρί συντονισμό οδήγησε σε χάο ε, αρχικά. Το καλό όμω είναι ότι βλέπουμε πόσο στενά συνδεδεμένοι είμαστε μεταξύ μα, όχι μόνο διασυνοριακά και όχι μόνο οικονομικά. Είδαμε ότι η ελευθερία μας είναι ευάλωτη, είναι πολύτιμη και θα πρέπει να την προστατεύσουμε. Ευτυχώς το Σέγγεν επανέρχεται στο σωστό δρόμο, η Ευρώπη επανέρχεται στο σωστό δρόμο και έχουμε πολύ δρόμο ακόμα μπροστά μας. Ας ε, Εξάγουμε λοιπόν τα λογικά συμπεράσματα. Α προετοιμάσουμε καλύτερα το Σέγγεν και να το εκμεταλλευτούμε στο έπακρον για την ανάκαμψη τη Ευρώπη. Α βγει η Ευρώπη πιο ισχυρή από όλα αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρο. Ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα το λόγο έχει η κυρία Τσιμέσκα. Για... Ο κύριο Τσιμέσκα, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, Επίτροπε. Θα μιλήσω αγγλικά. Στα σλοβακικά, συγγνώμη. Στη γλώσσα μου. Το Μάρτιο για πρώτη φορά αντιληφθήκαμε πόσο ευάλωτη είναι αυτή η ελευθερία μας. Αυτή η ελευθερία που λάβαμε χάρη στο χώρο Σέγγεν ήταν πραγματικά μια έκτακτη κατάσταση η οποία απαιτούσε προφανώς και έκτακτα μέτρα. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο τα κράτη-μέλη προέβησαν ε, στην ανάλυση δράσης, ε, χωρίς τονισμό δηλαδή, χωρίς νομικές βάσεις, όλα αυτά θεωρώ ότι ε, αποδυνάμωσαν την αμοιβαία εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Σέγγεν δεν είναι μια πολυτέλεια την οποία την ε, απολαμβάνουμε όταν ο καιρό είναι καλό. Είναι ο ακρογωνίος λίθος επί του οποίου βασίζεται η Ευρώπη μας. Δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι το πρώτο, η πρώτη αντίδραση, ακαρία αντίδραση των ευρωπαϊκών μελών είναι να κλείνουμε νούμερο στα σύνορά του. Θα πρέπει να εξαγάγουμε τα μαθήματα που χρειάζεται. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το Σέγγεν, ποιος θα είχε πιστέψει στην επιτυχία της συμφωνίας μιας μικρής πόλης που βρίσκεται σε παραμεθόρια περιοχή. Κι όμως ήταν το σύμβολο μιας Ευρώπης χωρίς σύνορα. Έγινε τόσο φυσική μετάβαση από τη μία χώρα στην άλλη που δεν μπορούσαμε καν να διανοηθούμε ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να σταματήσουμε και να δώσουμε δικαιολογητικά. Ήταν ένα ανεκτήμητο κεκτημένο λοιπόν το Σέγγεν. Ένα πραγματικό θαύμα τη Ευρωπαϊκή Ενότητα. Θα πρέπει να το διαφυλάξουμε αυτό το κεκτημένο. Η πανδημία COVID-19 σίγουρα δικαιολόγησε κάποιε περιορισμού μετακινήσει. Και η δημιουργία υγειονομικού κλειού όταν έχουμε πανδημία είναι φυσιολογικό. Ακόμη και τα σύνορα, η επαναφορά του μεταξύ χωρών μπορεί να είναι δικαιολογημένη κάποια στιγμή. Πώ όμω δικαιολογείται το κλείσιμο των σύνορων όταν έχουμε παρόμοια επιδημιολογική κατάσταση μεταξύ των γειτονικών χωρών. Είναι διανόητο σε μια στιγμή πανικού τα κράτη-μέλη να δράσουν με αναδίπλωση. Βέβαια, μπορεί να είναι φυσιολογικό κάτι και να εξηγείται, αλλά θα πρέπει το συντομότερο δυνατό τα κράτη-μέλη να ξανανοίξουν τα εσωτερικά του σύνορα στο χώρο Σέγγεν και να προετοιμαστούμε για την κρίση, γιατί δεν θα πρέπει να περιμένουμε μία έκτακτη περίπτωση για να ε, αναλάβουμε δράση. Διακόπτη δυστυχώ ο πρόεδρο ε, την ομιλήτρια. Σα ευχαριστώ, συνάδελφε. Ο κ. για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, η ελεύθερη διακίνηση για πάνω από 400 εκατομμύρια πολίτες είναι από τα θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βέβαια, όταν έχουμε μια πανδημία είναι κατανοητό ότι προσωρινά επαναφέρουμε τα εσωτερικά σύνορα. Η Ευρώπη όμως που γνωρίζουμε δεν νοείται χωρίς ελεύθερη διακίνηση των πολιτών. Αυτό είναι νευραλική σημασία και για την οικονομική ανάκαμψη και για τον τουρισμό αλλά και για τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωή. Χαίρομαι που το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δίνει ισχυρή υποστήριξη στην περαιτέρω διεύρυνση του Σέγγεν και στι υπόλοιπε τέσσερι χώρε μέλη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για την Κροατία, που είναι έτοιμη να αποτελέσει τμήμα του μεγαλύτερου χώρου ελεύθερη διακίνηση στον κόσμο, όπω δήλωσε πέρυσι και η πρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σήμερα είχαμε όμω ε, την ευκαιρία να ακούσουμε πάλι μια επίθεση κατά τη ε, χώρα μου ε, λόγω της ε, αποτελεσματικής πολιτικής προστασίας στα μεγαλύτερα χερσαία σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ελπίζω πολύ σύντομα και οι Κροάτες πολίτες, όπως και οι υπόλοιποι υπήκοοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να απολαύσουν το αγαθό της ελεύθερης διακίνησης και γι' αυτό χρειάζεται συνεργασία μεταξύ των κρατών μέλων και καλύτερη προστασία των εξωτερικών συνόρων. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και τώρα για ένα λεπτό ο συνάδελφος ο κ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε, αξιότιμη κυρία Επιτροπέ. Αν ε, είχατε ζήσει κι εσείς επί τρεις μήνες κοντά στα σύνορα, θα είχατε διαπιστώσει αυτοπροσώπως πόσο ε, καταπατήθηκε με πρωτοφανή τρόπο το Σέγγεν. Όταν σε τέτοιες εποχές κρίσης τα εθνικά κράτη-μέλη κλείνουν τα σύνορα χωρίς να έχουν μιλήσει μεταξύ τους δεν υπάρχει καμία επικοινωνία και δεν υπάρχει και καμία εμπιστοσύνη και τα δύο είναι πολύ άσχημα ούτε σε ό,τι αφορά το κλείσιμο των σύνορων ούτε στο άνοιγμα το σταδιακό διαφορών οικονομικών δραστηριοτήτων ούτε σε ό,τι αφορά την επανένωση οικογενειών υπήρξε συντονισμό, ούτε φυσικά σε ό,τι αφορά τη συνολική στρατηγική εξόδου. Αυτό οδήγησε λοιπόν ένα κατακριματισμό σε ό,τι αφορά όλα τα μέτρα. Κανείς δεν κατάλαβα τι έγινε, πώς θα μπορούσε άλλωστε. Για παράδειγμα, στο Βέλγιο ε, υποβάλαμε μια, ένα αίτημα για ε, σε μια νέα μορφή 2,0 προκειμένου αυτοί οι εθνικοί χώροι να καταστούν και πάλι κοινωτικοί χώροι. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει και ο πρόεδρος. Και τώρα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ακούσουμε την Επιτροπή Γιώχανσον. Thank you. Σας ευχαριστώ. Το Σέγγεν σημαίνει ελευθερία και βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη. Το Σέγγεν είναι μεγάλο επίτευγμα και αυτό φαίνεται και από την προσήλωση του Κοινοβουλίου στο θέμα αυτό και στην ε, επαναφορά μιας πλήρως λειτουργικής ζώνης Σέγγεν. Όταν ε, υπεγράφει αυτή η συμφωνία ε, πριν από 35 χρόνια, εκατομμύρια Ευρωπαίων ε, δεν είχαν δικαίωμα καν να εγκαταλείψουν τη χώρα τους. Τους τελευταίους μήνες θυμηθήκαμε ε, πώς ε, είναι η Ευρώπη χωρίς ελεύθερη κινητικότητα. Τώρα αργά και υπεύθυνα επανακτούμε τις ελευθερίες μας. Δεν μπορούμε να θεωρήσουμε δεδομένη την ελεύθερη κυκλοφορία, ούτε τα σημαντικά ωφέλη της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Κάθε μέρα πρέπει να εργαζόμαστε σκληρά για να προστατεύουμε και να διατηρούμε ε, τα ωφέλη του ευρωπαϊκού εγχειρήματος. Ε, καταρχάς, θα ήθελα να δω την απαραίτητη τη απόφαση του ε, Συμβουλίου για να μπορέσουμε να καλωσορίσουμε στη ζώνη Σέγγεν τα κράτη-μέλη που περιμένουν να μπουν. Αλλά θα πρέπει να κάνουμε κάτι καλύτερο από το να επανέλθουμε απλά στην, ε, στη συνηθισμένη κατάσταση των πραγμάτων όλες οι χώρες που θέλουν ε, να γίνουν μέλη της ζώνης Σέγγεν θα πρέπει να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα θεμελιώδη δικαιώματα και το ευρωπαϊκό κεκτημένο φυσικά. Ε, η ζώνη Σέγγεν βασίζεται σε αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών και στην σωστή εφαρμογή του κεκτημένου. Ε, ε, ε, γεγονότα σε ένα κράτος μέλος, ένα μπορούν να επηρεάσουν όλα τα άλλα κράτη και να διακυβεύσουν το μέλλον της ζώνης Σέγγεν. Θα πρέπει να φροντίσουμε να είναι κατάλληλο για να πετύχει τους στόχους μας το πλαίσιο της ζώνη Σέγγεν. Θα πρέπει να έχουμε σωστή εφαρμογή. Αυτό αφορά και τους εσωτερικού συνολικούς ελέγχους, τους αστυνομικούς ελέγχους, την σωστή τεχνολογία την ενισχυμένη διασυνοριακή συνεργασία ε, και, τις, ε, και την ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα στις διάφορες ε, αρχές επιβολής του νόμου. Θέλουμε να προτείνουμε επανεκκίνηση του διαλόγου με όλα τα κράτη-μέλη και τακτικούς πολιτικούς διαλόγους υψηλού επίπεδου και με το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Είμαι διατεθειμένη να συνεχίσω την αγαστή συνεργασία με όλους σας εδώ στο Κοινοβούλιο για να πετύχουμε το σημαντικό αυτό στόχο. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Επίτροπε. Η Υπουργό Πυρνιάκ, στο όνομα του Συμβουλίου, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για την συζήτηση αυτή. Τα θέματα που αφορούν τους εσωτερικούς συνοριακούς ελέγχους είναι απαραίτητες για τη, τη διατηρήση του κεκτημένου Σέγγεν. Γι' αυτό το Συμβούλιο προσλέπει στη στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να έχουμε μια νομικά σωστή και λειτουργική ε, εφαρμογή ε, της ζώνης Σέγγενη οι Υπουργοί αποφάσισαν στην τηλεδιάσκεψη της 15ης Ιουνίου να προχωρήσουν με τρόπο συντονισμένο ε, με βάση τις αρχές της αναλογικότητα ε, και της μη διάκρισης ε, και ακολουθώντας τις γραμμές που περιγράφονται στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ώστε να έχουμε τελικά άρση ε, των εσωτερικών συνολικών ελέγχων ε, και των ε, περιορισμών ταξιδιού μέχρι τις 15 Ιουνίου. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ. Έληξε η συζήτηση. Η ψηφοφορία θα πραγματοποιηθεί αύριο. Δύο ανακοινώσεις έχω ε, σχετικά με, τις επιτροπές, ε, την Επιτροπή Άγκρη. Δόθηκε χθε προθεσμία 24 ε, ωρών για την υποβολή αντιρρήσεων. Δεν έγινε αυτό και γι' αυτό οι συστάσεις θεωρείται ότι έχουν υιοθετηθεί και θα δημοσιευτούν. Επίσης θα ήθελα να σας ακοινώσω ότι χθε. ότι δεν έχει υπάρξει ε, κάποια αντίρρηση σχετικά με τη διόρθωση που ανακοινώθηκε χθε στι 3, άρα και αυτή εγκρίνεται. Επίση, όσον αφορά την ε, το επόμενο μας ε, θέμα είναι η ε, προστασία των ε, διασυνοριακών και εποχιακών εργαζομένων. Ξεκινάμε λοιπόν τη συζήτηση με δήλωση της Υπουργού Πρινιάξ από το Συμβούλιο. Παρακαλώ. Thank you. Σας ευχαριστώ. Αξιότιμη Ευρωβουλευτέ, κύριε Επίτροπε. Οι διασυνοριακοί και εποχιακοί εργαζόμενοι απασχολούνται στη γεωργία, τον τουρισμό, στη... στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όταν ε, δεν έχουν τα κρατημέρια αρκετά εργατικά χέρια. Είναι δύσκολο να δουλεύει κανείς μακριά από το σπίτι, οπότε θα πρέπει να προστατεύσουμε αυτούς του ευάλωτους εργαζόμενους ιδιαίτερα σε αυτούς τους πρωτοφανεί δύσκολους καιρού μετά το ξέσπασμα τη πανδημιας covid COVID-19. Τα μέτρα απομόνωση και κοινωνική αποστασιοποίηση είχαν ουσιαστικό αρνητικό αποτέλεσμα και επιζήμιο στην οικονομία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυξήθηκαν τα ποσοστά ανεργία πολύ σύντομα και οι επιχειρήσει αντιμετωπίζουν δυσκολίε σε μερικού τομεί πολύ περισσότερο από ό,τι σε άλλου. Τα κράτη-μέλη εφάρμοσαν ευρύ φάσμα μέτρων για να προλάβουν και να μετριάσουν σοβαρέ οικονομικέ επιπτώσει ε, στι αγορέ εργασία, στην κοινωνική ασφάλιση και το κράτο πρόνοια. Πολλά από τα μέτρα αυτά στόχο έχουν να προστατεύσουν του εργαζόμενου. Κυρίω σε ευαίσθητου τομεί και νευραλικού τομεί τη οικονομία. Και παρόλο που η υγειονομική έκτακτη ανάγκη υποχωρεί σιγά σιγά και τα μέτρα απομόνωσης περιοριστικά έρονται, οι οικονομικέ και κοινωνικέ συνέπειε παραμένουν σοβαρέ. Στι 5 Μαου, σε μια ε, τηλεδιάσκεψη που οργάνωσε η Κροατική Προεδρία, δώσαμε την ευκαιρία σε σε εμπλεκόμενους φορείς της κοινωνικής πολιτικής και της πολιτικής απασχόλησης να μας παρουσιάσουν τις απόψεις τους. Είναι σημαντική η προοπτική της κοινωνικής οικονομικής τη και οι υπουργοί τάχθηκαν υπέρ μια συντονισμένη προσέγγισης για να εξασφαλίσουμε απασχολησιμότητα, να στηρίξουμε τις επιχειρήσεις και να προστατεύσουμε του εργαζόμενου, κυρίω ε, του έχοντας ιδιαίτερα ανάγκη. Και μάλιστα το θέμα των συνοριακών και εποχιακών εργαζομένων προέκυψε πολλέ φορέ στη συζήτηση. Αυτή η ευάλωτη ομάδα είναι πολύ σημαντική για πολλού οικονομικού τομεί και θα παίξει ζωτικό ρόλο στην οικονομική ανάκαμψη. Και γι' αυτό θα πρέπει να υφίσταται διακριτική μεταχείριση τα μέλη αυτή τη ευάλωτη ομάδα. Η πανδημία COVID-19 ανάγκασε τα κράτη-μέλη να κλείσουν προσωρινά τα σύνορά του. Παρ' όλα αυτά, τα κράτη-μέλη και τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ε, δήλωσαν στην ε, κοινή τους διακήρυξη της 26ης Μαρτίου ότι ε, θα πρέπει να εξασφαλιστεί ομαλή διακίνηση αγαθών και πολιτών για την εύρυθμη λειτουργία της ευρωπαϊκής αγοράς. Και παρόλο που μερικά κράτη-μέλη ήραν τα περιοριστικά μέτρα για τη διακίνηση των διασυνοριακών και αποχιακών εργαζομένων, δεν το έχουν κάνει αυτό όλα τα κράτη-μέλη. Επίσης θα πρέπει να εξασφαλίσουμε αξιοπρεπεί όρου εργασία. Είναι το ίδιο σημαντικό με την ελεύθερη διακίνηση. Θα πρέπει να τη χάνουν ίσε μεταχείρισει αυτοί οι εργαζόμενοι. Παρόμοιε συνθήκε με αυτέ που ισχύουν για, τις, για του εργαζόμενου τη ίδια χώρα. Θα πρέπει επίσης ε, να έχουν κατάλληλο εξοπλισμό προστασίας ε, και κατάλληλες συνθήκες διαμονής με σεβασμό των μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης. Επίσης θα πρέπει να ενημερώνονται για τις αλλαγές και τις νέες διαδικασίες. Τα κράτη-μέλη επίσης δεσμεύτηκαν να εξασφαλίσουν πρόσβαση σε κοινωνική ασφάλιση, σε προσιτές τιμές σε όλους τους διασυνοριακούς εργαζομένους. Και η αναθεώρηση του κανονισμού για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης θα διευκολύνει περαιτέρω την ελεύθερη διακίνηση εργαζομένων και θα αποτελέσει καταλήτη στον εξυγχρονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γιατί κράτησε ε, ω σημαντική προτεραιότητα τα προβλήματα των συνοριακών και εποχιακών εργαζομένων και περιμένω με ανυπομονησία τη συζήτηση που θα ακολουθήσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την Υπουργό κυρία Κεμπρίνιατς και τώρα να ακούσουμε τον Επίτροπο Σμιτ. Πρόεδρε, αγαπητοί βουλευτέ η ελεύθερη μετακίνηση των εργαζομένων είναι βασική θεμελιώδης αρχή της Ευρωπαϊκής Ενιαίας Αγοράς. Εκατομμύρια Ευρωπαίοι ζουν και δουλεύουν σε άλλο κράτος μέλος από αυτό στο οποίο έχουν ε, υπηκότητα. Έχουμε μισό εκατομμύριο εποχιακούς εργαζόμενους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπολογίστητε. Και η κρίση γιατί με τον COVID-19 έχει οδηγήσει σε ανεφορεγμένου κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση με μεγάλο αντίκτυπο στην ελεύθερη μετακίνηση των εργαζομένων. Αυτό φάνηκε και στην προηγούμενη συζήτηση. Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι το εξής και είναι σαφής. Να εξασφαλίσει την ελεύθερη κυκλοφορία των ε, εργαζομένων. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, 30 Μαρτίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε κατευθυντήριε γραμμέ για την άσκηση του δικαιώματο αυτού τη ελεύθερη μετακίνηση από του εργαζόμενου. Σε ό,τι αφορά λοιπόν του διασυνοριακού και εποχιακού εργαζόμενου που ε, έχουν ε, κρίσιμε ε, θέσει να επιτελέσουν θα πρέπει να έχουν πρόσβαση χωρίς περιορισμό στις θέσεις τους αυτές. Και μιλάμε λοιπόν για εργαζόμενους και να σας πω ότι αυτοί οι εργαζόμενοι περιλαμβάνουν και πολλούς εποχιακούς εργαζόμενους που στην κρίση αυτή έχουν επιτελέσει ένα έργο πολύ σημαντικό και έχουν εργαστεί για κρίσιμα αγαθά και κρίσιμες υπηρεσίες. Τρόφιμα, για παράδειγμα. Για να εξασφαλίσουμε λοιπόν περαιτέρω σαφήνεια σε ό,τι αφορά το καθεστώ κοινωνική ασφάλεια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε και ένα φύλλο με ερωταπαντήσει με πληροφορίε για όλους τους διασυνοριακού και αποσπασμένου εργαζόμενου σε ό,τι αφορά ε, τα θέματα που άπτονταν της ελευθερίας μετακίνησης των COVID-19 βάσει στον διάλογο με τα κράτη-μέλη ξέρουμε ότι αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές είχαν θετικό αντίκτυπο. Συνεχίζουμε να παρακολουθούμε τα μέτρα τα οποία επιβάλλουν τα κράτη-μέλη, αν είναι αναλογικά και απαραίτητα για την καταπολέμηση του ιού και κατά πόσο δεν συνεπάγονται διακριτική μεταχείριση. Βασική τομή τη ευρωπαϊκής ε, οικονομία, ο γεωργικός και ο τουριστικό κλάδο κυρίω ε, ε, απαιτούν την υποστήριξη από εποχιακού εργαζόμενου για κάποιε περιόδου. και αυτοί οι εποχιακοί εργαζόμενοι συχνά είναι ευάλωτοι. Ευάλωτοι σε καταχρήσεις, σε επισφαλή συνθήκες εργασίας και συνθήκες διαβίωση, και σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στι δημόσιε υπηρεσίε και στη σωστή αξιοπρεπή στέγαση. Η παραβίαση λοιπόν του δικαίου σε ό,τι αφορά το καθεστώ ε, κοινωνικής ασφάλειας επίσης ε, συχνά είναι θύματα μη δηλωμένη ε, και μη καταχωρισμένη εργασίας. Η πανδημία COVID-19 θεωρώ ότι προέβαλε πιο πολύ και επέτεινε τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν πολλοί εποχιακοί εργαζόμενοι εδώ και πάρα πολύ καιρό. Η κατάσταση προσφάτως βελτιωνόταν. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν σοβαρά προβλήματα τα οποία εξακολουθούν να υπάρχουν για τους εποχιακούς εργαζόμενους και τα οποία θα πρέπει να επιληθούν. Η αρχή αυτή λοιπόν η οποία ισχύει για τους εποχιακούς εργαζόμενους είναι σαφέστατη. Ίση αντιμετώπιση και καμία διακριτική μεταγύριση των ε, εργαζομένων αυτών σε σχέση με τους εθνικούς εργαζομένους. Αυτό θα δώσει την καλύτερη δυνατή προστασία για τους εργαζομένους αυτούς που μετακινούνται και μεταξύ αυτών και τους δεσυνοριακούς και εποχιακούς εργαζόμενους. Για τους εποχιακούς εργαζόμενους τι σημαίνει αυτό, ότι έχουν τα ίδια ακριβώς δικαιώματα όπως και οι κάτοικοι του κράτους μέλους στο οποίο εργάζονται. Ίση αντιμετώπιση, ίση μεταχείριση σημαίνει τη σωστή εφαρμογή του εθνικού δικαίου και των νόμων αυτών που προκύπτουν από τις ευρωπαϊκές οδηγίες για τους εργαζόμενους που μετακινούνται. Δεδομένου ότι κάποιοι κλάδοι τη οικονομίας και κυρίως ο κλάδο της γεωργία προαπαιτεί την υποστήριξη από του εποχιακού εργαζόμενου από άλλα κράτη-μέλη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από τα κράτη-μέλη να ανταλλάξουν πληροφορίε και να δημιουργήσουν σαφεί ε, διαδικασίε για την ομαλή αντιμετώπιση των ε, εργαζομένων αυτών. ορίζω λοιπόν τη δήλωση που υπογράφτηκε στις 15 Μαΐου για τους εποχιακούς εργαζόμενους από τους Ευρωπαϊκούς Κοινωνικούς Εταίρους στον τομέα της Γεωργίας. Και επίσης καλώς ορίζω την ανακοίνωση των κρατών μελών να εγκρίνουν εθνική νομοθεσία και να ε, παρακολουθήσουν με καλύτερο τρόπο την εφαρμογή της. Τα δεδομένα μας ε, επιβεβαιώνουν ότι συχνά η δουλειά η εποχιακή δεν ε, δηλώνεται. Υπάρχουν καταχρήσεις σε ό,τι αφορά επίσης τη σωστή πρόσβαση στην κοινωνική πρόνοια. Άρα είναι απαραίτητο να ευαισθητοποιηθούν αμφότεροι εργοδότες και εργαζόμενοι σε ό,τι αφορά τα ωφέλη αλλά και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εποχιακοί εργαζόμενοι. Και αυτό είναι τμήμα της ε, σχετικής ε, εκστρατείας για την Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για την αντιμετώπιση της μη δηλωμένη εργασίας. Η Ευρώπη λοιπόν ε, εστιάζεται στις δραστηριότητες για τους δυσνοριακούς εργαζόμενους, τους εποχιακούς εργαζόμενου και κυρίω τους νέου στο εγγύησε μέλλον και η πλατφόρμα και το Ευρωπαϊκό Γραφείο Συντονισμού θα μεταφερθούν υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εργασίας, η οποία θα παρέχει αρρωγή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του κινητικού δικαίου, σε ό,τι αφορά την, ε, τους εργαζόμενους που μετακινούνται, και σε ό,τι αφορά την διακριτική μεταχείριση, αλλά και σε ό,τι αφορά τη σωστή πρόσβαση στη σύστημα κοινωνική πρόνοια. Ένα από του κανόνε σε ό,τι αφορά το συντονισμό αυτό είναι τα να εξασφαλίσουμε ότι τα άτομα τα οποία εργάζονται σε δύο και παραπάνω κρατημέλη, όπω οι εποχιακοί εργαζόμενοι, ακολουθούν το δίκαιο του κράτου μέλου με το οποίο έχουν του πιο στενού συνδέσμου. Προκειμένου να υπάρχει μια σταθερότητα και μια ασφάλεια στην πρόσβαση στα συστήματα κοινωνικής προστασίας, γιατί κάτι διαφορετικό θα αποτελούσε εμπόδιο για την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζόμενων. Είμαι βεβαισμένο ότι η αμοιβαία συνεργασία μεταξύ κρατών μελών, οι διμερεί συμφωνίε για παράδειγμα, ή για παράδειγμα η παροχή πληροφοριών στη γλώσσα των εποχιακών εργαζομένων, είναι απαραίτητα βήματα για να προστατευτούν τα δικαιώματα των ανθρώπων αυτών. Και η αναθεώρηση του σχετικού κανονισμού για την οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε πρόταση το 2016. Ακόμα βρίσκεται η υποφάση συζήτηση μεταξύ του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου και είμαι πραγματικά υπέρ της σωστής μεταρρύθμισης της νομοθεσίας και θα ήθελα να υποστηρίξω την εισαγωγή ενός ευρωπαϊκού α, κοινωνικού μητρώου. Να πω και κάτι άλλο. Δεδομένη τη κρίση ανευπροηγουμένων την οποία διανύουμε, πρόκειται για ένα ζήτημα στο οποίο δεν μπορούμε να αποτύχουμε. Δεν μπορούμε να εγκαταλείξουμε τους πολίτες μας. Θα πρέπει το σύστημα αυτό να ισχύει για όλους τους πολίτες, ανεξάρτητα από το που δουλεύουν, ε, τη διάρκεια ή τη φύση της εργασίας που επιτελούν η εξασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων είναι κοινή μας ευθύνη. Είναι ευθύνη των εργοδοτών να εκπληρώνουν όλες τις ε, προδιαγραφές για όλους τους κινδύνους στον χώρο εργασίας, συμπεριλαμβανομένων και των νέων κινδύνων και να εφαρμόσουν σωστά και κατάλληλα και δέοντα μέτρα προστασίας. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα σε κλάδους όπου ενδεχομένω να έχουν μεγάλη έκθεση οι εργαζόμενοι. Οι εργοδότε επίση υποχρεούνται να παρέχουν σωστέ πληροφορίε προς τους εργαζόμενους, καθώς και το σωστό προστατευτικό εξοπλισμό και εξοπλισμό υγιεινής. Πέρα από τις κατευθυντήριε γραμμέ για τους εποχιακούς ε, εργαζόμενους και την σχετική προετοιμασία, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει λάβει πολλά βήματα για να υποστηρίξει τους, ε, τα κράτη-μέλη Προ την κατεύθυνση αυτή. Θέλω να προσθέσω το εξή όμως. Τα κράτη-μέλη έχουν ευθύνη να ελέγχουν την εφαρμογή των ε, εργατικών δικαιωμάτων που ισχύουν φυσικά και για τους εποχιακούς ε, εργαζομένους. Η Ευρωπαϊκή όσα δημοσίευσε ε, κατευθυντήριες γραμμές για την αντιμετώπιση του COVID-19 στο χώρο εργασία, καθώς και σχετικά με την ε, ασφαλή επιστροφή στο χώρο εργασία μετά τον COVID. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τις πτυχές για την ε, ασφάλεια και την υγεία, γίνεται αναφορά και στις εθνικές ε, νομοθεσίες. Ιδιαίτερα για τους κλάδους εκείνους που χρησιμοποιούν πολλούς εποχιακούς εργαζόμενους και σας διαβεβαιώ ότι η προστασία των εργαζομένων αυτών και τη υγεία και τη ασφάλειά του θα είναι βασική προτεραιότητα τα επόμενα χρόνια και θα συνεργαστώ στενά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να ενημερώσω και το στρατηγικό πλαίσιο του ισχύ και να κοιτάξουμε τις συνέπειες σε ό,τι αφορά την υγεία και την ασφάλεια του COVID και σε ό,τι αφορά τους πιο ευάλωτους εργαζομένους. Δεν ξεχνάμε ότι πολλοί εποχιακοί εργαζόμενοι είναι και πολίτες τρίτων χωρών και η κρίση COVID-19 είχε σημαντικό αντίκτυπο στη δυνατότητα να μπουν, να εισέλθουν στην Ένωση οι άνθρωποι αυτοί. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι αυτοί οι εργαζόμενοι, ιδιαίτερα στον κλάδο της γεωργίας, συχνά επιτελούν σημαντικό έργο. Και γι' αυτό λοιπόν το Μάρτιο ζητήσαμε από τα κράτη-μέλη να εγκρίνουν την ε, είσοδο των εργαζομένων αυτών τρίτων χωρών στον τομέα της γεωργίας παρά το κλείσιμο των συνόρων. Και καλώς ορίζω λοιπόν το ψηφίσμα σας ως μια σημαντική συμβολή για την κατάρτιση μιας μελλοντικής πολιτικής. Θέλουμε να πετύχουμε το ίδιο στόχο, να εξασφαλίσουμε ότι τα δικαιώματα των εποχιακών εργαζομένων προστατεύονται και ότι εφαρμόζονται οι κοινοτικοί κανόνες και ότι όλα αυτά ισχύουν για όλους. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε, ο συνάδελφος Λέναρς. Ευχαριστώ πρόεδρε. Συχνά οι λαϊκιστές εδώ στην Κοινοβούλιο λένε ότι θα πρέπει να φύγει το Σέγγεν και να κλείσουν τα σύνορα. Αυτή είναι η εικόνα ε, που προβάλλουν και αυτή ήταν δυστυχώ η εικόνα που ζήσαμε τους τελευταίους μήνες και αυτό ε, το σενάριο του Βίλτερ της Λεπέν και ε, πολλών άλλων ε, είναι ένα σενάριο εφιαλτικό για εκατομμύρια πολίτες που ζουν κοντά στους, ε, στα σύνορα που βλέπουν τις καλλιέργειές τους, τις παράγκε τους, τις φράουλες τους να σαπίζουν γιατί κανείς δεν μπορεί να τα μαζέψει για τους επιχειρηματίες σε διασυνοριακό επίπεδο που βλέπουν τις επιχειρήσεις τους να μαραζώνουν και διαπιστώνουμε λοιπόν πόσο σημαντικά είναι όλα αυτά. Και είναι σημαντικό αυτό το μάθημα που πρέπει να εξαγάγουμε. Να μην μπούμε σε την παγίδα αυτή του ας κλείσουμε τα σύνορα, ας ε, ε, προστατεύσουμε την αγορά εργασίας μας και μια δυσνοριακή εργασία, αγορά εργασίας, όπου η αξιοπρεπής διαβίωση είναι ο κανόνας και που προστατεύονται τα δικαιώματα όλων και δεν επικρατεί η κακή πίστη. Αυτή είναι η δική μου το δικό μου σενάριο για το μέλλον της Ευρώπης. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Μπίσοφ, ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χθες στην Γερμανία βρήκαμε εκατοντάδες νέα περιστατικά κοροναϊού σε μια μεγάλη κρεατοβιομηχανία. Αυτό εμένα μου δείχνει ότι κανένας δεν έμαθε τίποτα από την κρίση και ότι ε, με ανευθυνότητα προχωράμε και ε, προσπαθούμε να ρίξουμε το φταίξιμο στους ε, φτωχούς Ρουμάνους εργαζομένους επειδή έφεραν διασυνοριακά τον ιό. Δεν επιτρέπεται να συμβαίνει κάτι τέτοιο, δεν επιτρέπεται να δώσουμε χώρο στον λαϊκισμό, γι' αυτό χρειάζεται ακριβώς ένα τέτοιο ψήφισμα. Πρέπει να βελτιώσουμε την Ευρώπη εκεί που υπάρχουν ελλείψεις και θα πρέπει να ε, φροντίσουμε για την καλύτερη εφαρμογή του δικαίου. Θα ήθελα όμως να κάνω και μία έκκληση προς όλους ε, τους ε, εποχιακά και διασυνοριακά εργαζομένους. Σας παρακαλούμε μην χάσετε τις ελπίδες σας για μια ελεύθερη και δίκαιη αγορά εργασίας ε, στην Ευρώπη. Εμείς ε, εδώ στο Κοινοβούλιο συνεχίζουμε να καταβάλουμε προσπάθειες με στόχο αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Τσιόλος. Κύριε Επιτροπέ, αγαπητοί συνάδελφοι, Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να εντοπίσουμε το αντικείμενο αυτού του ψηφίσματος. Οι διασυνοριακοί και εποχιακοί εργαζόμενοι είναι αυτοί που ε, δίνουν πνοή ζωή σε πολλούς οικονομικούς κλάδους. Πρόκειται για πολλούς πολίτες που αφήνουν τις αισθήσεις και τις οικογένειές τους για αρκετά μεγάλη περίοδο από τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία για παράδειγμα και πηγαίνουν στην άλλη γωνιά της Ευρώπης για να βοηθήσουν την οικονομία σε άλλα κράτη-μέλη. Και αυτοί οι άνθρωποι στέλνουν χρήματα στις οικογένειές τους, στα παιδιά τους που έμειναν στην πατρίδα τους. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε ένα ολόκληρο κλάδο Τη Ευρωπαϊκή οικονομία που εξαρτάται από αυτού του εργαζόμενου. Η κρίση μα έδειξε ότι αυτοί οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να κινηθούν ελεύθερα ε, και να περάσουν τα σύνορα. Έτσι κινδυνεύει ολόκληρη η παραγωγή, ε, όπως κινδύνευσαν ε, οι μεταφορές, ο τουρισμός, ή η παροχή φροντίδα και υγειονομική περίθαλψη. Είναι σημαντικό να αντιληφθούμε τη σημασία που έχουν οι εργαζόμενοι αυτοί για την ευρωπαϊκή οικονομία και για τα κράτη-μέλη. Για τη γεωργία, για παράδειγμα, ή για τα νοσοκομεία για τον κατασκευαστικό οικοδομικό κλάδο και για πολλούς άλλους τομείς. Θα πρέπει λοιπόν να προστατεύσουμε αυτούς τους εργαζόμενους. Αυτό είναι το ελάχιστο καθήκον που θα πρέπει να αναλάβουμε, γιατί χωρίς τους εργαζόμενους αυτούς πολλοί νευραλγικοί κλάδοι της οικονομίας θα κινητοποιηθούν. Διαπιστώσαμε με την κρίση ότι πολλοί εποχιακοί εργαζόμενοι διαμένουν σε άθλιες συνθήκες διαμονής, χωρίς καν να στοιχειώδη υγιεινή και όταν ασθενούν δεν έχουν καν πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας. Μερικοί αρρωσταίνουν, πεθαίνουν ε, και δεν μπορούν να απολαύσουν τα κοινωνικά τους δικαιώματα. Η ομάδα Renew λοιπόν ε, πρωτοστάτησε στην σύνταξη αυτού του ψηφίσματος που στηρίζεται από μεγάλη πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θέλουμε να σεβαστούμε τα δικαιώματα αυτών των εποχιακών εργαζομένων που αξίζουν αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης και αξιοπρεπείς αμοιβέ. Δεν θα πρέπει να τους ε, τιμωρούμε γιατί ήδη είναι τα θύματα αυτή τη κατάσταση. Θα πρέπει λοιπόν να συνεργαστούμε με τα κράτη-μέλη, την Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να ε, του βοηθήσουμε σε αυτού του δύσκολου καιρού. Η κυρία Ζαμέ για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, το ψήφισμα αυτό που ρυθμίζει την ελεύθερη ε, διακίνηση και την προστασία των εργαζομένων, άσχετα με το καθεστώ του, δημιουργεί πρόβλημα. Για μία ακόμη φορά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να κατοχυρώσει τον ιερό και απαράβατο χαρακτήρα τη ελεύθερη διακίνηση των εργαζομένων και άρα τη απόσπαση των εργαζομένων. Ε, Επίση, μιλά για την ε, ισότιμη μεταχείριση και την αποφύγη των διακρίσεων που αντιβαίνουν στι εθνικέ προοπτικέ και προτεραιότητε όμω που μα είναι ιδιαίτερα προσφυλή. Στην ίδια κατηγορία βάλουμε του διασυνοριακού, του εποχιακού και του αποσπασμένου εργαζομένου. Αυτό είναι απαράδεκτο. Άλλωστε το κείμενο αυτό αντιβαίνει στα θεμελιώδη και ζωτικά συμφέροντα των συμπολιτών μα. Θα πρέπει να διαγράψουμε του αποσπασμένου τους αποσπασμένους εργαζομένους στην απόσπαση εργασία και να προωθήσουμε τι εθνικέ προτεραιότητε. Σα ευχαριστώ. Η κυρία έχει τώρα το λόγο. Κυρία Υπουργέ, Πρόεδρε, Επιτροπέ, αυτή η πανδημία α, σημαίνει επισφαλής θέση εργασίας για 17 εκατομμύρια άτομα. Χρειαζόταν ήδη καλύτερη προστασία η ομάδα αυτή πριν από την κρίση, αλλά η έλλειψη προστατευτικών μέτρων σε ό,τι αφορά α, ε, τους εργαζόμενους στα σφαγεία και στα χωράφια φράουλα στην Ολλανδία και στη Γερμανία άνοιξαν τα μάτια όλων γιατί οι προδιαγραφές ε, υγείας και ασφάλειας για τον COVID-19 δεν τηρούνται πάντα και η... το πέρασμα των σύνορων θα πρέπει να είναι καλύτερα, θα είναι πιο εύκολο για αυτούς και θα πρέπει να υπάρξει επίσης καλύτερο συντονισμός. Αυτό είναι κατεπήγον. Αυτοί οι άνθρωποι είναι στην πρώτη γραμμή, στα νοσοκομεία για παράδειγμα στην Αυστρία, όπου έχουμε πολλούς, ε, πολλές νοσοκόμες για παράδειγμα από τη Ρουμανία οι οποίες επιτελούν σημαντικό έργο. Θα πρέπει να φροντίσουμε την απαραίτητη κοινωνική προστασία και την προστασία της ε, εργασίας και της υγείας και της ασφάλειας των ανθρώπων αυτών. Είναι θέμα κοινωνικής δικαιοσύνης. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Ντεσίτερ. Και τώρα η κυρία Ραφάλσκα για ένα λεπτό. Κύριε Επίτροπε, αξιότιμοι συνάδελφοι. Οι διασυνορικοί και εποχιακοί εργαζόμενοι ε, επλήγησαν ε, ιδιαίτερως από την πανδημία COVID-19 λόγω των κλειστών συνόρων, των περιοριστικών μέτρων και της καραντίνας και ενίοτε αδυνατώντα να επιστρέψουν στη χώρα τους ή να λάβουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ή να έχουν και μέσα βιοπορισμού. Περισσότερο από άλλους εργαζόμενους λοιπόν εξαρτάται εξαρτώνται από τους εργοδότες και τις, τα γραφεία ανέβρης εργασίας. Οι συνθήκε διαμονής τους είναι άθλιες μερικές φορές, υπολείπονται κάθε προδιαγραφές και έχουν πολύ χαμηλές αμοιβέ και επίσης πολύ χαμηλές προδιαγραφές ασφάλειας και υγιεινής. Όλα αυτά δείχνουν τι τεράστια προβλήματα αντιμετωπίζουν οι διασυνοριακοί και εποχιακοί εργαζόμενοι που πολύ συχνά προέρχονται από την Ανατολική Ευρώπη. Η πανδημία μάλιστα κατέδειξε πόσο απαραίτητοι και υποτιμημένοι είναι αυτοί οι εργαζόμενοι, από του οποίου εξαρτώνται πολλοί κλάδοι τη οικονομία. Θα πρέπει λοιπόν να αναγνωρίσουμε την αξία του, να οριθετήσουμε ε, σωστέ συνθήκε εργασία γιατί ε, και πριν την πανδημία υπήρχαν πολλές καταχρήσεις ε, εις βάρος των εργαζομένων αυτών Το σκέφτηκε καθόλου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τι μέτρα θα λάβει. Δυστυχώς διακόπτει ο Πρόεδρος. Κυρία συνάδελφε, δεν μπορούμε να υπερβαίνουμε έτσι το χρόνο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ένα λεπτό, συνάδελφος Μποτέγκα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, θα ψηφίσουμε ένα ψηφίσμα για τα δικαιώματα των, εργασία... των εποχιακών, αποσπασμένων και διασυνοριακών εργαζομένων. Και χαίρομαι ιδιαίτερος που συμμετείχα στη σύνταξη αυτή, όχι μόνο με την αριστερή παράταξη, αλλά και με τους φιλελεύθερους και τη δεξιά παράταξη. Και είναι πραγματικά καταπληκτικό που για πρώτη φορά αναγνωρίζουμε ότι η απόλυτη προτεραιότητα στην αγορά βλάπτει τα δικαιώματα των εργαζομένων. Ξέρω ότι δεν είστε έτοιμοι να μιλήσετε για κοινωνικό ντάμπινγκ. Αν είστε έτοιμοι, πολύ ευχαριστώ να σα υποβάλω σχετική τροπολογία για να την υπερψηφίσετε. Θα σα ενθαρρύνω πάντω και θα χαιρετήσω και θα χειροκροτήσω το ψήφισμα που θα υιοθετήσουμε σήμερα. Η πανδημία κορώνα 19 μας άνοιξε τα μάτια στα δεινά των διασυνοριακών και ε, εποχιακών εργαζομένων λέτε. Δεν σας πιστεύω. Νομίζω ότι η πίεση που νιώσατε είναι αυτή που σας άνοιξε τα μάτια. Είδατε πόσο ε, αντικείμενα εκμετάλλευση γίνονται αυτοί οι εργαζόμενοι που ε, συνοστίζονται μερικές φορές σε μεγάλα φορτηγά και βρίσκονται σε άθλιες συνθήκες διαμονής και εργασιακέ. Αυτό που με ενδιαφέρει όμω είναι πώ θα συνεχίσουμε από εδώ και πέρα. Γιατί το ψήφισμά μα δεν είναι δεσμευτικό πολύ καλά που θα το ψηφίσουμε και θα το εγκρίνουμε, αλλά θα πρέπει να κάνουμε και ένα βήμα ακόμη και θα πρέπει να προσαρμόσουμε του ευρωπαϊκού κανόνε και διατάξει, ώστε τα δικαιώματα των εργαζομένων πραγματικά να υπερτερούν έναντι των οικονομικών ελευθεριών και να επικρατούν έναντι τη αγορά. Σα ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ένα λεπτό η κυρία Ροντινέλη. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η πανδημία μας έχει δείξει αυτές τις εβδομάδες ότι η ευρωπαϊκή αγορά είναι πολύ πιο ολοκληρωμένη από ό,τι φανταζόμασταν. Αντιληφθήκαμε ότι χωρίς την ελεύθερη διακίνηση των εργαζομένων και κυρίως των εποχιακών και διασυνοριακών εργαζομένων, ολόκληρη παραγωγική στρατηγική τομή της οικονομίας κινδυνεύουν να κινητοποιηθούν ο εργαζόμενο, όταν αφήνει την πατρίδα του, την ε, χώρα προέλευσής του μέσω του πράσινου διαδρόμου, θα πρέπει να τύχει προστασία με υψηλέ προδιαγραφές ε, και αξιοπρεπεί προδιαγραφές διαμονής, ε, εργασία και αμοιβή και να ληφθούν υπόψη και τα κεκτημένα του και τα κοινωνικά δικαιώματα που θα πρέπει να επιβαρύνει το η χώρα που εργάζεται ο εργαζόμενο και εκεί που πληρώνει του φόρου. Θα πρέπει λοιπόν να προωθήσουμε την εναρμόνιση των εθνικών εργασιακών νομοθεσιών, να διορθώσουμε το εργασιακό dumping και το μισθολογικό dumping και να αποφύγουμε και το dumping στην υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Μπορούμε να ε, θα υιοθετήσουμε το ψήφισμα και ελπίζω να αποτελέσει τη βάση για νέε νομοθετικέ διατάξει για να εξασφαλίσουμε καλύτερη προστασία των Ευρωπαίων εργαζομένων και να αποφύγουμε τον αθέμητο ανταγωνισμό που δυστυχώ μαστίζει ακόμη την ενιαία ευρωπαϊκή αγορά. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ, ο κύριος Ράτκε. Κύριε Πρόεδρε, συνάδελφοι. Συστημική είναι Συστημικός είναι η λέξη που είναι της μόδας ε, και ε, αναφέρομαι ε, τώρα στην σημασία της ελεύθερης κινητικότητας και των ελευθεριών, αλλά βλέπουμε τώρα και πόσο βάλλοντο είναι το σύστημα αυτό. Τσέχοι νοσοκόμοι που εργάζονται στη Γερμανία έπρεπε από τη μία μέρα στην άλλη να αποφασίσουν να διαλέξουν ανάμεσα στην οικογένειά τους ή τη δουλειά τους και αγρότες ε, ξαφνικά είχαν πρόβλημα με την ε, συγκομιδή τους και στον ε, τομέα του κρέατος στα σφαγεία της Γερμανίας πάλι είδαμε σημαντικά προβλήματα. Γι' αυτό είναι θετικό ότι το Κοινοβούλιο υποβάλλει αυτό το ψήφισμα και να αναπόκειται πια στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προχωρήσει σε πράξεις. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Δύο λεπτά η κυρία Γιονγκέριος. Ευχαριστώ πρόεδρο. Διαρωτάται κανείς. Τι σκέφτεται κανείς όταν ε, από την Πολωνία τη Ρουμανία έχει έρθει για να δουλέψει 14 ώρες την ημέρα, 42 μέρες συνεχόμενες συναπτές. Τι ε, μπορεί να σκέφτεται κάποιος που θέλει να τον πετάξει στον δρόμο τον άνθρωπο αυτό, τον, αυτό το μετανάστη, γιατί έχει απλά πυρετό και τον παρατάει στην άκρη του δρόμου και τον αφήνει στην τύχη του σε μια ξένη χώρα. Αυτά δυστυχώς είναι παραδείγματα από τη χώρα μου, την Ολλανδία, την τελευταία εβδομάδα. Θα σκέφτονταν ε, κανείς, μα τι μπορεί να σκέφτεται αυτός ο άνθρωπο. Δεν μπορεί κανείς να πετάει στον δρόμο τους ανθρώπους. Δεν είναι σκουπίδια οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι. Ε, ο γεωργικός κλάδος και ο κλάδος παραγωγής τροφίμων έχει καταρρεύσει και από Δύση μέχρι Ανατολή όλοι συμφωνούμε ότι κάτι θα πρέπει να γίνει και θα πρέπει να υποβάλουμε προτάσεις για να αντιμετωπίσουμε τις καταχρώσεις αυτές. Ε, να υπάρχουν δεσμευτικοί κανόνες ε, με ενημέρωση της σχετικής οδηγίας για τους Αποσπασμένου, ε, ζητήματα αντιμετώπισης της στέγασης των ανθρώπων αυτών με privacy και επίσης ε, εποπτεία και παρακολούθηση της στήριξης των προδιαγραφών αυτών με επιθεωρητές. Περιμένω από εσά, Επίτροπε Σμιτ, να αντιμετωπίσετε άμεσα τα προβλήματα και τι καταχρήσει που διαπιστώνουμε και να ε, προωθήσετε το ψήφισμα αυτό. Τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να υποβάλουν μέτρα, θα πρέπει να αναλάβουν δράση. Γιατί το να δουλεύει κανείς σε μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα είναι δικαίωμα των εργαζομένων αλλά θα πρέπει όλοι να μπορούν να είναι βέβαιοι ότι είναι ασφαλές το περιβάλλον εργασίας τους. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Την κυρία Γιονγκέριος. Τώρα για ένα λεπτό το λόγο έχει ο κύριος Πισλάρου. Το ψήφισμα της ομάδας Ρινιού που είχα την τιμή να συντονίσω και όλα αφιερώνεται στους ε, Ρουμάνους, Βούλγαρους, Πολωνούς, συνοριακούς και παχιακούς εργαζομένους. Ε, αποτείουμε φόρο τιμής ε, σε εργαζόμενους που υπέσαν τεράστια προβλήματα. Μερικές φορές έχασαν και τη ζωή τους, συνοστισμένοι σε εμπορευματοκιβώτια ή σε φορτηγά στην προσπάθειά τους να βοηθήσουν την ευρωπαϊκή οικονομία. Η κρίση αυτή δεν είναι καινούρια ε, στους κλάδους αυτούς. Οι εποχιακοί εργαζόμενοι είναι ένα σύμβολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμβολο της ε, ευημερίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σύμβολο της εσωτερικής αγοράς. Εμείς λοιπόν είπαμε να αφογκραστούμε τις ανάγκες αυτών των εποχιακών και διασυνοριακών εργαζομένων και να δώσουμε μάχη για να γίνουν σεβαστά τα δικαιώματά τους, τα δικαιώματα των εργαζομένων παντού στην Ευρώπη. Δικαίωμα σε αξιοπρεπείς ε, συνθήκες εργασίας και διαβίωσης. Έχουμε το ηθικό καθήκον να, να μεριμνήσουμε για τους ανθρώπους αυτούς τώρα και στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ συνάδελφε. Ε, ο κύριος Πάνσα, ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Με κάποιες επιφυλάξεις ε, μπορώ να συμφωνήσω με το ψήφισμα αυτό. Ε, για την η περίπτωση της Ιταλίας ε, μιλάμε για πάνω από 100.000 ε, διασυνοριακούς εργαζόμενους που εργάζονται για παράδειγμα στη Γαλλία ή στο Σαν Μαρίνο και 17.000 στην Ελβετία. Πρέπει λοιπόν ε, να φροντίσουμε να έχουν ε, ε, ανθρώπινες συνθήκες εργασίας και να προστατέψουμε όλους τους διασυνοριακούς εργαζομένους. Τα κράτη-μέλη λοιπόν πρέπει να εφαρμόσουν κατάλληλα μέτρα. Θα πρέπει να φροντίσουμε επίσης να υπάρξει νομοποίηση των παρανόμως εργαζομένων. Αυτό έγινε στην Ιταλία και επίσης πρέπει να υπάρχουν νόμοι μέσοδοι μετανάστευση. Σας ευχαριστώ πολύ. Για ένα λεπτό, Σατούρη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, με την κρίση του COVID-19, τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ευθύνονται για πολλές παραβιάσεις των δικαιωμάτων των ε, μετακινούμενων εργαζομένων. Με την απότομη, με το απότομο κλείσιμο των συνόρων, οι πιο ευάλωτοι από τους εργαζόμενους, κυρίως από ε, τρίτες χώρες, έμειναν μόνοι και ανήμποροι, ανυπεράσπιστοι απέναντι στις καταχρήσεις των εργοδοτών τους, χωρίς πόρους, σε άθλιες συνθήκες διαβίωσης, χωρίς καν τη δυνατότητα μερικές φορές να επιτρέψουν στις πατρίδες τους Ό,τι και να λένε οι εθνικιστέ, αυτοί οι άνθρωποι έχουν ουσιώδη σημασία για την οικονομία μα, για τη γεωργία μα, για την ανοικοδόμηση των χωρών μα. Και πραγματικά η μεταχείριση που του επιφυλάσσουμε είναι ανάξια των ευρωπαϊκών αξιών. Η ισότητα των δικαιωμάτων θα πρέπει να κατοχυρωθεί για όλους γιατί θεωρητικά υπάρχει, αλλά θα πρέπει να κάνουμε ένα ακόμη βήμα. Ήρθε η ώρα να περάσει η Ευρώπη από την εκμετάλλευση των μεταναστών εργαζομένων στην αναγνώριση της συμβολής του στην οικονομία μας και στην ε, επισητιστική μας κυριαρχία. Θα πρέπει η ισότητα των δικαιωμάτων να γίνει πραγματικότητα απτή και ε, επαληθεύσιμη. Σας ευχαριστώ. Και τώρα η ε, κυρία Νίκολσον για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε 1,3 διασυνοριακού εργαζόμενου και 2 εκατομμύρια αποσπασμένου εργαζόμενου. Στην κρίση COVID-19 διαπιστώσαμε πώ ε, ευάλωτοι είναι αυτοί οι εργαζόμενοι. Και όταν ε, κλείνουν τα σύνορα, αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να επιλέξουν κατά πόσον θα μείνουν κοντά στην οικογένειά του και δεν θα εργαστούν ή θα εργαστούν και θα μείνουν χωρισμένοι από την οικογένειά του. Και έτσι λοιπόν ε, ο τομέα τη κοινωνική προστασία, ο τομέα τη γεωργία, ο τομέα των μεταφορών έμειναν ε, με μεγάλη έλεψη προσωπικού και έτσι συχνά βλέπουμε στα κοινωνικά συστήματα να υπάρχουν μεγάλες διατάξει διακριτική μεταχείριση, για παράδειγμα στην Αυστρία, σε ό,τι αφορά τα οικογενειακά επιδόματα. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει συντονιστό των κοινωνικών ε, συστημάτων και να υπάρχει ψηφιακή σύνδεση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Ντούρι Νίκολσονοβά και τώρα η κυρία Σάιμπη έχει το λόγο για ένα λεπτό. Αγαπητοί συνάδελφοι, καλημέρα. Θα ήθελα να σα μιλήσω για τη Γιασμίνη. Γιασμίν που μαζεύει ε, φρούτα, τα πεπόνια, τα ροδάκινα που μας αρέσουν και τις δίνουν ψίχουλα κάθε μήνα της Γιασμίν. Όταν ε, ε, θέλει να φάει δεν έχει δικαίωμα να κάνει διάλειμμα και πρέπει να τρώει στα κρυφά στις τουαλέτες και πάσχει και από μια σοβαρή νευρολογική ασθένεια και αυτό είναι η πραγματικότητα των εκατοντάδων αποσπασμένων εργαζομένων, εποχιακών εργαζομένων, οι οποίοι έρχονται από την Ισπανία και σε κάποιε περιπτώσει είναι από τη Γουινέα, από την Κολομβία, που έχουν αποσπαστεί στην Γαλλία, τη Γερμανία ή και αλλού για να μαζέψουν φρούτα και λαχανικά. Η κρίση του COVID-19 προέβαλε όλες αυτές τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν αυτοί οι εργαζόμενοι τους οποίους ε, υπόκονται καταχρήσεις σε ε, ακραίες συνθήκες μάλιστα λόγω της εξάπλωσης του COVID-19. Η κατάχρηση αυτών των ανθρώπων θα πρέπει να σταματήσει των γυναικών και των ανδρών. Είναι απαράδεκτη και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εξασφαλίσει τα δικαιώματα των ανθρώπων αυτών μέσω τη οδηγία για του αποσπασμένου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Κυρία Σάιμπη, λέει ο Πρόεδρος, δεν βλέπω να είναι στην αίθουσα ο κύριος Ραντασόφσκι. Άρα το λόγο παίρνει ο κύριος Μπούντα για ένα λεπτό.